Il eh, Καλησπέρα σε όλους. Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης είναι πλέον διαθέσιμα. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι. Επομένως εγκρίνονται τα πρακτικά. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε κοινή συζήτηση για